Συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στην ε, από κοινού συνεδρίαση με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, στήριξη για έκτακτες ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποδοχή των ετούντων άσυλο στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη το 2015 στην Ελλάδα όπου πέρασαν πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ερχόμενοι από τον πόλεμο στη Συρία και από, άλλους, από άλλες περιοχές, Όλοι γνωρίζουν πως η Επιτροπή Ντεβε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του στήριξε τη χώρα αυτή, διασφαλίζοντας ότι θα υπήρχαν χρημα... κονδύλια και χρηματοδότηση ΕΚΟ για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτό ήταν κάτι το άνευ προηγουμένου, να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα ανθρωπιστικής ε, βοήθειας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό δημιουργήθηκε και το ESI, το Emergency Support Instrument, που σε 200 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί στην UNICEF σε διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στην αρμόδια αρμοστία των Εθνών για τους πρόσφυγες και σε άλλους φορείς για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν και άλλα ε, κονδύλια που είναι διαθέσιμα. Ο Πολ Μωράης θα μας πει περισσότερα, ο Κλοντ Μωράης θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Όμως, στα τέλη Ιουλίου, οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη για το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, της δουλειάς που μέχρι αυτή τη στιγμή κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι διεθνείς οργανώσεις. Οι ελληνικές αρχές θα αρχίσουν οι ίδιες να τρέχουν τα προγράμματα και ο σκοπός μας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο θα είναι ομαλή αυτή η μετάβαση μεταξύ της δουλειάς της χρηματοδότησης ΕΚΟ, της χρηματοδότησης ανθρωπιστικής βοήθειας και της χρηματοδότησης που ε, θα περάσει πλέον στις ελληνικές αρχές για να ε, κάνουν όλες αυτές τις υπηρεσίες ε, σε σχέση με τους ετούντες άσυλο στην Ελλάδα. Δυστυχώς ο Έλληνας Υπουργός δεν μπόρεσε να έρθει εδώ, ο κύριος Μουζάλας, και δεν έχουμε εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης σήμερα το πρωί. Λυπούμε γι' αυτό. Έχουμε όμως εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να δώσω το λόγο στον κύριο Κλοντ Μωράες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Λίντα. Χαίρομαι ιδιαίτερως διότι συνεδριάζουν από κοινού οι δύο αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να εξετάσουμε τη μεταβατική περίοδο της χρηματοδότησης του ΕΚΟ η οποία απευθυνόταν στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε άλλους φορείς και τώρα πλέον θα περνάει από τις ελληνικές αρχές. Έχουμε επισκεφθεί επί τόπου την κατάσταση. Ε, θελήσαμε να ευχαριστήσουμε και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που μας διευκόλυναν σε αυτό το καθήκον και είχαμε την ευκαιρία και να συλλέξουμε διάφορες πληροφορίες. Άρα αυτά που κάνουμε σήμερα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δική μας ανάλυση, στη βοήθεια που είχαμε από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους ανεξάρτητους συνομιλητές και διαλειτουργικούς συνομιλητές. Σκοπός της σημερινή συνεδρίασης νομίζω ότι είναι να εξετάσουμε τα διάφορα έργα που ε, χρηματοδοτούνται από το σχετικό ταμείο της ελληνικής κυβέρνησης και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το, από το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σταδιακή εξάλληψη χρηματοδότησης από το Emergency Fund, από το Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτοκτων Καταστάσεων και είχαμε τις σοκαριστικές εκθέσεις τον περασμένο χειμώνα για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά, τις οποίες γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε συνεχιζόμενες αφήξεις, ακόμα και αν τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την υποδοχή των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι θα συνεχίσει να υπάρχει εξασφάλιση και εγγύηση γι' αυτό. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουμε πρόσωπο. δυστυχώς από πλευράς ελληνικών αρχών δεν έχουμε, δεν μπόρεσε ο Έλληνας Υπουργός να παραβρεθεί. Θα ακούσουμε όμως από την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες για τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο αλληλεγγύης με την Ελλάδα. Πρέπει να αναλύσουμε ποια θα είναι η κατάσταση εφ' εξής. Επομένως, ο ομιλητής θα μας χαρτογραφήσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο Σάιμον Μόρτζι, αναπληρωτής γενικός διευθυντής, ο οποίος έχει έρθει πολύ συχνά να μας δει το τελευταίο στάδιο, το τελευταίο καιρό και θα μας μιλήσει για αυτή τη μετάβαση. Σάιμον, να σας δώσουμε το λόγο για 7-8 λεπτά. Ο Σάιμον Μόρτζι, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω όλοι γνωρίζετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που ανατρέχει τον Οκτώβριο του 2015. Στην κορύφωση της κρίσης είχαμε χιλιάδες μεταναστών που έφταναν και πώς να βρουν τη διαδρομή των δυστικών Βαλκανίων. Υπήρχαν μεταβίες 2.000 θέσεις για όλη τη χώρα και δεν ήταν καλέ οι συνθήκε υποδοχή, αλλά ούτε οι δυνατότητε ούτω ώστε να υπάρξει κάποιο είδου καταγραφή ε, και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων για αυτού του μετανάστε. Ε, και αν ήταν εδώ ο κύριο Μουζάλα, θα τον επενούσα για τι συνεχεί του προσπάθειες και ακάματε όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ακόμα υπάρχουν κάποιε προκλήσει, αλλά η κατάσταση έχει σημαντικά βελτιωθεί. Και αυτό διότι έχουν γίνει συνεννοημένε προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων, όχι μόνο των ελληνικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνεί οργανώσεις, κοινωνία των πολιτών, όλοι με τον τρόπο τους συνέβαλαν τόσο ώστε να υπάρξει πρόοδο. Και από πλευρά μα ως Επιτροπή, ε, να σας πω συγκεκριμένα τι έκανε η ΕΚΟ, κινητοποίησαμε ό,τι μέσα υπάρχουν εμπειρογνωμοσύνη και ε, χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ε, για την μετανάστευση και να γίνουν όλα μας με πιο ανθρωπιστικό τρόπο. Ξεκινούμε για το θέμα της χρηματοδότησης γιατί έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι ε, με το ISF και AMEF και αυτά ξεκινούν το 2014 μέχρι το 2020 Και από αυτά τα προγράμματα 509 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν αυτών όμως από την αρχή της μεταναστευτικής κρίσης κινητοποίησαμε 362 εκατομμύρια, τα οποία ήταν κάτι σαν κατεπίγουσα αρρωγή, είτε άμεσα στις ελληνικές αρχές ή μέσω ε, του IOM, άλλων οργανώσεων όπως την τη αρμοστία του ΟΗΕ. Και πρόκειται λοιπόν για μια έκτακτη κινητοποίηση αυτής της επιπλέον χρηματοδότησης και αυτά τα είδαμε να πιάνουν από κάθε μέρα με τις ομάδες μας, με τον ε, Μάρτιν στην Αθήνα και ήταν τρομερή η καθημερινή συνεργασία με τις ελληνικές ε, αρχές. Ε, επίσης αναπτύξαμε και κάποιους ειδικού από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου, από την Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή, όλα αυτά για να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές. Αυτό που θέλω τώρα να σας αναφέρω είναι ότι πρόκειται για μια σαφή απόδειξη της αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις η Ελλάδα, να μπορέσει να κάνει κάτι για αυτή την τεράστια μεταναστευτική πίεση. Και αυτά τα συζητήσαμε ε, προηγουμένως με το θέμα του διαδρόμου της κεντρικής ε, Μεσογείου και είπαμε ότι θα πρέπει η υποστήριξη να προσφερθεί αελεγγύη από τα κράτη-μέλη και αυτό να είναι βιώσιμο. Αλλά πρόοδο δεν είδαμε στο Συμβούλιο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου. Και επίσης σε αυτό όλο το ψηφιδωτό λείπουν πολλά κομμάτια. Δεν έχει βρεθεί βιώσιμη λύση για αυτά τα προβλήματα με τον Πεζή Ελλάδα. Δύο λόγια τώρα όσον αφορά ε, τι σχέσεις με την Τουρκία και τη σχετική δήλωση. Δεν έχουμε ε, τα αποτελέσματα. Ε, πέραν του ότι έχουν πέσει σημαντικά οι αφήξεις στην Ελλάδα, επίσης ε, μειώθηκαν ε, οι απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Οπότε, να, τώρα υπάρχει καλύτερο έλεγχο των σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα οι μετανάστες και οι ετούντε άσυλο επίση έχουν μειωθεί. Ακόμα υπάρχουν προκλήσει, η κατάσταση είναι πιο ανθρώπινη για την υποδοχή αλλά θα πρέπει να τονίσουμε, θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, να εξομαλυνθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιες δυσκολίες στην ε, χείο, σχετικούς καταβλισμούς και επομένως θα πρέπει πηγόντως κάτι να κάνει η Ελλάδα και από πλευρά μα έχουμε εντείνει προσπάθειες για βελτίωση των συνθήκων μία από τις ήταν και γι' αυτό είπαμε να βοηθήσουμε με τρόπο βιώσιμο και γι' αυτό και ήρθαμε σε επαφή, συνεργασία με την Ελλάδα για αυτό που θέλουμε να γίνει το 2017 προγραμματισμός ούτως ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να γίνει πιο καλή χρήση της χρηματοδότησης που ήδη έχει διατεθεί προς την ε, χώρα για τα εθνικά προγράμματα επομένως τώρα θέλουμε οι ευρωπαϊκές αρχές να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να γίνει μια ταχεία υλοποίηση αυτού του προγραμματισμού έχουν ε, αναβαθμίσει προσπαθιές τους για αξιοποίηση αυτών των κοινωτικών χρημάτων με αυτά τα πολιτή εθνικά προγράμματα και αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε να δούμε πώς εθνικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν ούτως ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής των μεταναστών και πιο συγκεκριμένα βλέπουμε με ικανοποίηση ότι τώρα έχουν ε, ε, γίνει σχετικοί διαγωνισμοί για την υποδοχή στα νησιά και αξιολογούνται αυτές οι προσφορές και τώρα ε, υπάρχει διαδικασία πρόβλεψης για κάποιους καταβλισμούς για ασυνόδευτους ανηλίκους και έχουν γίνει από το Υπουργείο τις τελευταίες εβδομάδες σημαντικές προσπάθειες. Είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε αυτό το θέμα των συνόθων ανηλίκων γιατί αυτοί είναι η πιο ευάλωτοι και αυτοί θα πρέπει ε, σε κάθε ε, εγκατάσταση να προσέχονται. Επίσης γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν προβληματιστεί για αυτό που λένε ότι είναι η μη συνεχιζόμενη οικονομική βοήθεια προς τα νησιά. Ξεκαθαρίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η οικονομική βοήθεια διοχετεύεται από διαφορετικούς διάβλους, δηλαδή από τα εθνικά προγράμματα και η διαχείριση και η εποπτεία γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα θα συνεχίσουμε να δερματίζουμε κάποιον ρόλο σε αυτή τη μετάβαση και ο Ζων θα σας πει τις λεπτομέρειες για την δουλειά της ΕΚΟ. Συνεχίζουμε και φροντίζουμε για διάφορα κέντρα υποδοχής αλλά ακόμα είναι τεράστιες οι ανάγκες και ένα από αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και οπότε τώρα τα εθνικά προγράμματα έχουν ακόμη περισσότερη χρηματοδότηση μια προσέγγιση να έχουμε που θα την ονόμαζα ως αντίδραση βιώσιμη. Το νωρίτερο που θα ε, φύγουμε από αυτή την κατάσταση κατεπίγουσας διαχείρισης όπου έχει βοηθήσει αποτελεσματικά ο στρατός σε κάποιο είδους ε, διαχείριση κατά την οποία οι, οι υπηρεσίες ε, παρέχονται βιώσιμα από τα εθνικά θεσμικά όργανα. Αυτό θα ωφελήσει τους πάντες. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά την ποιότητα των συνθήκων υποδοχής. Προσπαθούμε επομένω να προχωρήσουμε, να μην υπάρχει υποδοχή μόνο σε αυτά τα στρατούς καταβλισμούς τους προσωρινούς, αλλά να είναι σε άλλα μέρη πιο μόνιμα, πιο ε, αξιοπρεπή. Να μην έχουμε τις ε, σκηνές ε, των οποίων γίναμε μάρτυρες το χειμώνα, τα Χριστούγεννα πέρσι. Άρα, ούτε αφέθηκε μόνη της η Ελλάδα, ούτε θα αφαιθεί. Εμείς θα συνεχίσουμε ε, δραστήριοι να βοηθούμε με αυτήν την οικονομικό προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός ε, επιδέχεται και πρόκειται να προσαρμοστεί όπως χρειάζεται. Θα βοηθήσουμε τις αρχές, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε στενόμυαλοι. Να, παράδειγμα, έχουμε... Ε, μια αποστολή της ε, βουλευτών της ΛΥΜΠΕ στην Λέσβο στο Καρατεπέ και εκεί ε, τα πράγματα ήταν πολύ συμπαθητικά, οικογενειακά αλλά υπήρχαν ε, δυσκολίες για τη συνεχή παροχή της οικονομικής βοήθειας αλλά τώρα υπάρχει πρόγραμμα ούτως ώστε να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών στο Καρατεπέ και όταν πήγα εκεί μου εξήγησε ο Δήμαρχος για το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και είπαμε ότι υπάρχει θέμα με τα διευθυντικά ταμεία και με τον Επίτροπο βρήκαμε ε, κάποια λύση ούτως ώστε αυτό το, αυτό το δαπάνες αυτές να υποστηριχθούν. Άρα δείξαμε την ευελιξία ε, για το κόστος και για το πόσο ε, ανοιχτόκαρδα οι κάτοικοι του νησιού βοήθησαν. Δηλαδή και με την καλύτερη δυνατή διαχείριση και προγραμματισμό δεν μπορεί όλα να γίνουν από το βράδυ ως το πρωί. Οπότε και όλο τον ε, Αύγουστο θα είμαστε έτοιμοι, θα έχουμε ομάδες ε, για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση είτε εδώ είτε όπως τα συζητήσαμε για τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου για εκεί. Άλλαν. Ευχαριστούμε, οπότε αυτό ήταν μια πρόγευση των όσων κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Με τον Κλοντ πήγαμε στο Καρατεπέ, συνδύσαμε και τον Δήμαρχο, που ανησυχούν όλοι για τον προπολογισμό και όλοι χρειάζονται υποστήριξη. Χαίρομαι πολύ για τις λύσεις που έχουν βρεθεί. Θα δώσουμε το λόγο και στον Ζωνίτη από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν κενά στη χρηματοδότηση μπορεί να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά σήμερα έχουμε 12 Ιουλίου και στο τέλος του μήνα θα περάσουμε στη νέα χρηματοδότηση. Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο από τις ελληνικές αρχές. Θέλουμε να δούμε, θα υπάρχουν υπηρεσίες, θα λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες την 1η Αυγούστου μετά τη μετάβαση γιατί αυτοί που λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν θα πρέπει ξαφνικά να καταλάβουν ότι υπάρχει διαφορά. Η υπηρεσία πρέπει να συνεχίσει να παρέχεται ακόμη και αν αλλάξει το κανάλι χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας για τη μετάβαση αυτή και για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που μόλις είπε ο Σάιμον Μότζιου. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα τα έχουμε εντοπίσει και οι περισσότερες λύσεις έχουν ήδη βρεθεί. Παρουσίασα στην Επιτροπή σας την πρώτη ετήσια έκθεσή μας τον Απρίλιο και σας είχα πει τότε ότι υπάρχουν κάποιοι άξονες εξέλιξης για την κοινή δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες ειδικές μας και οι υπηρεσίες του Σάιμον. το χρηματοδοτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε από τις ελληνικές αρχές και που εγκρίθηκε από τους δύο αρμόδιους επιτρόπους, τον Επίτροπο Στυλιανίδη και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, βασίζεται όσον αφορά τις υπηρεσίες του Επιτρόπου Στυλιανίδη στην συγκέντρωση των δράσεών μας στην υπηρετική Ελλάδα, και η διάρθρωση της παρέμβασής μας ε, βασίζεται στα δύο μεγάλα ε, μέσα που είναι ένα ε, πρόγραμμα παροχής μετρητών και όπως έλεγε ο Σάιμον προοδευτική ανάπτυξη ενός συστήματος καταλημάτων για τους πρόσφυγες. Ε, κάποια, κάποιοι χώροι έχουν τεθεί στη διάθεσή τους και τώρα που μιλάμε έχουν εγκαινιαστεί νέα καταλήματα με πολύ βελτιωμένες υποδομές. Η Αναμπέλ θα μπορέσει να σας πει περισσότερα για τον τρόπο εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων και για τους εταίρους ε, σε αυτή την προσπάθεια και μέχρι τα τέλη του έτους, ανάλογα με τις ανάγκες, θα διατεθούν νέα καταλήμματα. Τα βασικά ζητήματα είναι η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ε, και ο καλός συντονισμός. Ο συντονισμός εξ αρχής ήταν τέλειος μεταξύ των δύο δικών μας υπηρεσιών και σε βασικό επίπεδο στις Βρυξέλλες και επιτόπου διότι έχουμε και μια ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων επιτόπου στην Αθήνα. Και όπως έλεγε και ο Σάιμον, θα από την εξαιρετική υποστήριξη της υπηρεσίας του Μάρτιν Φέρβε που βρίσκεται επιτόπου στην Αθήνα και μαζί με τη δική μας ομάδα μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη αυτή και κατά την ε, ευαίσθητη αυτή μεταβατική περίοδο που αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα. Πρώτον, οι μη συνοδευόμενοι ανήλικοι και δεύτερον, το πέρασμα σε νέες πηγές χρηματοδότησης στα νησιά, όπως ανέφερε ο Σάιμον Μότζι. Όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, έχουμε σχετικά καλά νέα έγινε μια προκήρυξη για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση θέσεων για συνόδευτους ανηλίκους αντίστοιχος αριθμός όπως αυτές που έχουμε μέχρι σήμερα με υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων μία διαφορά κάποιων εκατοντάδων θέσεων ίσως να υπάρχει και την επόμενη εβδομάδα θα πάω στην Αθήνα και μαζί με τις ελληνικές αρχές θα διερευνήσουμε τους τρόπους ε, για να καλύψουμε αυτό το μικρό κενό. Μια καινούργια προκήρυξη προβλέπεται ήδη από ό,τι έχω ακούσει και αν γίνει εξίσου αποτελεσματικά όπως και οι προηγούμενοι ελπίζω ότι γρήγορα θα λυθούν οποιαδήποτε προβλήματα εάν υπάρξουν. Όσον αφορά τα νησιά, συμφωνώ με αυτά που έλεγε ο Σάιμον και πιστεύω ότι πρέπει να, τονίσουμε ότι ε, η παρέμβασή μας ήταν οριακή στα νησιά. Δεν είχαμε ποτέ ε, μαζική παρέμβαση από πλευράς ε, του ESI. 2.000 θέσεις σε καταλήμματα για τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες και συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε ε, κάποια μετρητά στα νησιά συμπληρωματικά με αυτά τα οποία μέχρι τώρα γίνονται. Η χρηματοδότηση θα είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ μέσω των διαφόρων έργων τα οποία χρηματοδοτούμε μαζί με τις υπηρεσίες του Σάιμον και με τους άλλους εταίρους μας θα συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε ε, κάποια χρηματοδότηση κατά αυτή τη μεταβατική περίοδο και την επόμενη εβδομάδα, όπως σας είπα στην επίσκεψή μου στην Αθήνα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση το συντομότερο δυνατόν. Δυστυχώ δεν είναι εδώ ο Υπουργό, ο κ. Μουζάλα, ε, που παίζει ένα ρόλο κλειδί, όπω είπε και ο Σάιμον, στο συντονισμό αυτής ε, της προσπάθειας σήμερα. Αλλά η έγκριση και η υλοποίηση ε, αυτού του προγράμματος χρηματοδότησης το 2017 μας επέτρεψε να βελτιώσουμε σημαντικά το συντονισμό και τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, κυρίως μέσω της παρακολούθησης των έργων, και της ανταπόκρισης στα αιτήματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι εταίροι μας. Όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων που αντιμετωπίσαμε και οι δύο υπηρεσίες το 2016, μπορούμε σαφώς να πούμε ότι έχει βελτιωθεί ε, κατά πολύ το κλίμα. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν, ευρώ δόθηκαν το 2016-2017 μέσω του ESI, του Emergency Support Instrument και άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ παραμένουν μέχρι το τέλος του έτους και για το 2018 δεσμευόμαστε για το τελευταίο έτος υλοποίησης ε, του χρηματοδοτικού κονδυλίου που μας δόθηκε από τη Δημοσιονομική Αρχή. Ήταν 300, 200 και 200 εκατομμύρια, τρεις δόσεις και κατά το επόμενο έτος θα είμαστε στο έτος ε, εξόδου συγγνώμη, από το ESI. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπογιέρ. Έχουμε μιλητή από την ε, ΥΠΑΤΗ Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και θα σας δώσω το λόγο. Είδα την πολύ καλή δουλειά που έχετε κάνει. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ρόικ. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που καλέσατε το UNHCR με, σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπως είπε και η Γενική Διεύθυνση HOME και η ECO, Πάρα πολλά χρήματα έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και εμείς έχουμε λάβει σε μεγάλο βαθμό αυτά τα κονδύλια με πλήρη διαφάνεια. Το 2015 και 2016 το UNHCR έχει λάβει περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ, 123 εκατομμύρια από την Γενική Διεύθυνση Home και 160 εκατομμύρια από την DG ECO για την ανθρωπιστική βοήθεια. Μεγάλα τα ποσά. περισσότερο από ό,τι έχει λάβει οποιαδήποτε άλλη χώρα ή υπηρεσία. Η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες με την ανταπάντηση που δίνει στην προσφυγική κρίση και συγκεκριμένα στα νησιά. Όλοι όμως συμφωνούμε ότι δεν είμαστε σε φάση επίγουσας αντιμετώπισης πια. Ε, έχουμε ενίσχυση των θεσμών, ενίσχυση των δεξιοτήτων επιτόπου και βιωσιμότητα. Αυτά μας ενδιαφέρουν αυτά μας ενδιαφέρουν, δεν, είναι, δεν χαρακτηρίζεται πλέον η κατάσταση ως απολύτως επίγουσα. Αυξάνονται τα αιτήματα ασύλου που υποβάλλονται στην Ελλάδα, αυξάνονται ο αριθμός των ανθρώπων που τους δίδεται διεθνής προστασία, δηλαδή το καθεστώς του πρόσφυγα ή κάτι άλλο και που ε, ε, κατ' επέκταση θα παραμείνει στην Ελλάδα. Ένα, μια επόμενη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή είναι η ανάγκη να έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκλήρωσης, ενοποίησης, integration program και αυτό θα είναι μια νέα θεσμική ε, πρόκληση, ε, ένταξης δηλαδή και πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα προγράμματα ένταξης και ενσωμάτωσης. Αυξάνεται το ποσοστό των αναγνωρίσεων και περισσότεροι άνθρωποι θα μείνουν στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι οι επενδύσεις στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου στην Ελλάδα για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα προχωρούν. 2.700 άνθρωποι πήραν το καθεστώς του πρόσφυγα πέρσι στην Ελλάδα και τους το αναγνωρίστηκε αυτό και φέτος άνω των 3.000 ατόμων θα τους αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα. Αυτή δεν είναι επιλέξιμη για μετεγκατάσταση, για relocation και θα πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα. Λίγες χιλιάδες ανθρώπων θα χρειαστούν περισσότερο μακροπρόθεσμες προοπτικές στην Ελλάδα. Όλοι αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της Ελλάδας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ελληνικός πληθυσμός. Θεωρούμε όμως ότι αυτά τα νούμερα νούμερα των 3.000 ανθρώπων που τελικά θα χρειαστούν κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση δεν είναι υψηλά νούμερα και είναι διαχειρίσιμα. Και ε, θεωρούμε ότι ε, πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος χρόνου. Επομένως το UNHCR το modus operandi το έχει αλλάξει στην Ελλάδα. Δεν είμαστε πια σε emergency, σε επίγουσα κατάσταση, αλλά σε post-emergency, σε μετά την επίγουσα κατάσταση. Στηρίζουμε τις κρατικές αρχές, τοπικές, εθνικές, να ε, εμπλακούν περισσότερο στο σύστημα ασύλου και να υπάρξει και η συνιστόσα της ενσωμάτωσης και της ένταξης των ατόμων ε, στους οποίους αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα. Έχει αυξηθεί η συνεργασία μας με τις δημοτικές αρχές, με τους δήμους, με τις τοπικές κοινότητες. Υπάρχει ανάγκη να συνεργαζόμαστε. Ορισμένες, ε, ορισμένοι δήμοι ήταν πραγματικά πάρα πολύ θετικοί στην ανταπόκρισή τους και συνεργάστηκαν εξαιρετικά καλά. Ένα παράδειγμα είναι ο Δήμος του Πειραιά, όπου έχουμε ένα πρόγραμμα υποδοχής, accommodation, καταλήμματων τα περισσότερα διαμερίσματα διαχειρίζονται οι μη κυβερνητικέ οργανώσει κατά κύριο λόγο ελληνικέ ΜΚΟ και ο Δήμο Πειραιά έχει συμφωνήσει να αναλάβει τη διαχείριση και τη λειτουργία 50 διαμερισμάτων τα οποία λειτουργούσαν πριν μη κυβερνητικέ οργανώσει. Μιλούμε δηλαδή για μια ένταξη, για μια ενσωμάτωση, για μια τέτοιου είδου διαδικασία που έχουν αναλάβει οι τοπικές αρχές, κάτι το επενεταίο. Είναι μια νέα επικοδομητική δυναμική και συνεργαζόμαστε με την ΕΚΟ, τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, για να τη στηρίξουμε. Ω σύσταση προτείνουμε να αυξηθεί η δημοποίηση, το twinning, μεταξύ ε, ελληνικών πόλεων και ε, άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, να γίνουν περισσότερες αδελφοποιήσεις πόλεων για να στηρίξει η μία την άλλη. πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους Δήμους που έχουν την πολιτική βούληση να συνεργαστούν και να ε, κάνουν το πάντα για να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση αυτών που θα μείνουν στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση στα, στα κονδύλια που είναι βάση της νομοθεσίας ΑΜΙΦ, ε, ε, δηλαδή χρηματοδότηση για θέματα ασύλου, μετανάστευσης και του καθεξής και ένταξης από το AMIF, Asylum Migration και Integration Fund και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές εκεί. Τώρα έχουμε δύο προγράμματα, ένα πρόγραμμα ε, καταλημάτων με στόχο τους ανθρώπους που θα μετεγκατασταθούν εκτός Ελλάδας. Αυτό σταδιακά άνοιξε και ε, περιέλαβε και τους ετούντες άσυλο και τώρα θέλουμε το ίδιο πρόγραμμα να στοχεύσει και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ένα δεύτερο πρόγραμμα, όπως είπε ο είναι το πρόγραμμα με ρευστό, με χρήματα. Βήματα για να αυξηθεί η αυτάρκεια των ατόμων και η ενσωμάτωσή τους και η ένταξή τους. Είναι μια πρόκληση αυτά να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Προωνίας για να είναι βιώσιμα μέσω μακροπρόθεσμα. Στηρίζουμε το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι εθνικοί φάκελοι να αξιοποιηθούν στο μέγιστο, στο πλαίσιο του Ταμείου για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη και την ενσωμάτωση και θα πρέπει η, τα, επίγουσα, τα επίγοντα κονδύλια σταδιακά να μειώνονται. Θέλουμε ε, ο στόχος ε, για τον εθνικό φάκελο να περιλάβει τις ανάγκες ένταξης και ενσωμάτωσης, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση, εκμάθηση της γλώσσας, ενίσχυση των συνδικών εργασίας των ανθρώπων αυτών. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, πολύ λεπτό ζήτημα. Είμαστε σε αυτή τη μεταβατική φάση αυτή τη στιγμή και από την κατεπίγουσα χρηματοδότηση προχωράμε στην αξιοποίηση των εθνικών προγραμμάτων και κονδυλίων και πρέπει αυτό να γίνει υπεύθυνα, με υπεύθυνο τρόπο, για να αποφύγουμε τον αρκτικό αντίκτυπο για τους ενδιαφερόμενους. Έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι ευαίσθητη αυτή η περίοδος του καλοκαιριού και θέλουμε να μην υπάρξουν κενά σε αυτή τη μεταβατική φάση. Ας πούμε θα, ε, στη διαχείριση που γίνεται των καταλημάτων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους ή για την παροχή υπηρεσιών στα νησιά, ε, στα κέντρα υποδοχής. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πως ο στόχος του προγράμματος υποδοχής ε, καταλημάτων δηλαδή 30.000 ατόμων στην επιρετική χώρα θα χρηματοδοτηθεί με επαρκή κονδύλια άπαξ και αφαιρέσουμε τα κονδύλια της κατεπίγουσας χρηματοδότησης ΕΚΟ. Ε, αυτό είναι κάτι που προβλέπεται για το ε, 2019, να έχει ήδη ολοκληρωθεί. Να κάνω ένα σχόλιο για την παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ στο ελληνικό τοπίο από πέρσι. Ήταν ένα ενδιαφέρον αυτός ο αστερισμός, αν θέλετε, πολλών και διαφορετικών παραγόντων που παρανέβηκαν στην Ελλάδα. Η ΕΚΟ είναι ένας ανθρωπιστικός παραγόντας με μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό. Αντιμετωπίσε πολύ μεγάλες προκλήσεις προσπαθώντας να δουλέψει σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην οποία οι κρατικές αρχές δεν μπορούν να παρακαμφθούν σε σύγκριση με άλλες ε, περιοχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν κάλεστα να παρακαμφθούν οι εθνικές κρατικές αρχές. Υπάρχει το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, κοινοί κανόνες και κοινό πλαίσιο. Όλα αυτά περιέπλεξαν την εργασία της ΕΚΟ, ήταν θέματα συντονισμού και συνεργασίας, κάτι το οποίο ε, δεν ήταν τόσο προφανές και τόσο εύκολο τα διαφορετικά και παράλληλα συστήματα να μπορέσουν να συνεργαστούν, δημιουργήθηκαν πολύ γρήγορα και, τα, ε, και εμείς ε, συμβάλαμε σε αυτό το μηχανισμό το συντονιστικό μαζί με τις ελληνικές αρχές, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω. Επίσης, ίσως είναι εξαιρετικά νωρίς για την αξιολόγηση του αντικτύπου της ΕΚΟ στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, ίσως μπορούμε να πούμε ότι πράγματι βγαίνει το εξής συμπέρασμα. Η εφαρμογή μιας στάνταρ ανθρωπιστικής προσέγγισης δεν μπορεί να ισχύσει εντός ενός κράτους μέλος και υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από αυτό. Τώρα, μελλοντικά, εμείς διαδραματίζουμε κρίσιμο ρόλο σε όλες τις πτυχές του ζητήματος των προσφύγων. Έχουμε το πρόγραμμα με το ρευστό και το πρόγραμμα με τα καταλήματα. Ε, δίνουμε, προσφέρουμε μετάφραση, διερμηνία, μεταφορές, νομική βοήθεια, προστασία ανηλίκων και το καθεξής. Σας έδωσα τα νούμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί κυρίως τη δουλειά μας, είτε η Γενική Διεύθυνση Home, είτε η Γενική Διεύθυνση ECO και είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε και να απεμπλακούμε από την Ελλάδα στο βαθμό που ε, αυτοί που θα πάρουν την σκητάλη το πράξουν με ε, υπεύθυνο τρόπο δεν μιλούμε για καλύτερες προβλέψεις, αλλά για περισσότερες προβλέψεις για το πώς θα προχωρήσουμε του χρόνου και του παραχρόνου. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που ήδη γίνεται και οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει για το 2018. Σε ό,τι μας αφορά θα πρέπει να είναι καλύτερες οι προβλέψεις μας για το πώς θα διαχειριστούμε τη στρατηγική εξόδου της ΕΚΟ, πώς θα διαχειριστούμε τη στρατηγική ε, της δικής μας μείωσης, της δικής μας παρέμβασης και πώς θα αυξηθεί το κομμάτι που αναλαμβάνουν οι ελληνικές κρατικές αρχές. Ο κύριος Μωράης, σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ε, προβλέψει να έχουμε τον Υπουργό μαζί μας για να του διαβιβάσουμε τις απόψεις μας. Αυτός είναι και ο σκοπός μιας έκτακτης συνεδρίασης. Εγώ τον συνάντησα στην Παρασκευή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και του μετέφερα τα βασικά που θα συζητούσαμε σήμερα το πρωί για τη μεταβατική αυτή περίοδο. Επομένω, έτσι, έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε τον Υπουργό μαζί μα. Όμω, σα καλώ να πάρετε το λόγο για να καταγραφούν οι απόψει σα και να τι μεταφέρουμε στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό. Ε, στρέφομαι λοιπόν προς τα μέλη των δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών για να τους δώσω το λόγο. Ξεκινούμε με τον Ενρίκε Γκερέρο, συντάκτη της εισηγήσης της έκθεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ, Κλοντ. Λέω ο κύριος Γκερέρο. Ναι. Και εγώ μαζί με άλλους ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία όσον αφορά το θεματολόγιο της Επιτροπής Ανάπτυξης και στη συνέχεια μέσα από την ΛΥΜΠΕ. Γιατί θέλαμε να επιδείξουμε ελληνική προς την ελληνική κυβέρνηση για τις προσπάθειες που κατέβαλε και επίσης προσπαθήσαμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που είχαν και τι είδους βοήθεια μπορούσαμε να παράσχουμε από δική μας πλευράς σαν κοινοβούλιο και από τα άλλα θεσμικά όργανα. Κρίμα που δεν είναι εδώ ο υπουργό. Αλλά έχουμε πλήρη ενημέρωση από τους τρεις ε, εισηγητές. Και θα ήθελα να ρωτήσω τα εξή και να παρατηρήσω κάτι. Τότε που είχαμε πάει σε ένα καταβλισμό κοντά στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Μουζάλα και αυτός ο καταβλισμός ήταν της τελευταίας γενιάς. Καλές οι συνθήκες. Ήταν ε, τέλη Μαρτίου, ήδη είχε περάσει ο χειμώνας και τα προβλήματά του, αυτά που ξέρουμε για την προηγούμενη χρονιά και ήταν προφανώς ότι τελείωσε η φάση της κατεπίγουσας ανάγκης και ότι άρχιζε η φάση του ότι θα έπρεπε με ε, εξομάλυνση να συνεχίσουμε όσον αφορά πρόσφυγες και μετανάστες. Ήδη επομένω είχε ξεκινήσει τουλάχιστον εκεί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην υπηρετική Ελλάδα, το πρόγραμμα της ε, μίσθωσης κατοικιών, ούτως ώστε να μεταφερθούν οι πρόσφυγες από τους καταβλισμούς σε εκείνα τα διαμερίσματα. Και είχα και έχω ακόμα την εντύπωση ότι υποσυνείδητα οι ελληνικές αρχές ακόμα αισθάνονται κάποια ανασφάλεια ότι ανά πάσα στιγμή η Τουρκία θα κάνει στροφή. Θα αλλάξει γνώμη και αφού φτάσαμε στη φάση της εξομάλυνσης, ότι ξαφνικά θα ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση της έκτακτης ανάγκης. Έτσι που συμπεριφέρονται αυτοί, αυτοί που είναι απέναντι από το Αιγαίο. Οπότε είπαμε ότι δημιουργείται αυτό το αίσθημα ανασφάλειας στις ελληνικές αρχές εν μέρη κατανοητό. Οπότε και αυτό ζημιώνει τις προσπάθειες, τις προσπάθειες σταθεροποίησης πλήρους της καταστάσεως. Ισχύει ότι δεν είμαστε σε κατάσταση δεκτά της ανάγκης, αλλά όπως μας είπε η κυρία Ρόχ, Γνωζόν, συγγνώμη, Ρότς, Ρότς, Ρότς είναι το σωστό. είναι Βέρα Βαλενθιάνα. Οπότε χρειάζεται ειδικέ γλωσσικέ γνώσει. Η σωστή προφράτονομα, το όνομα. Τόσα κύριε ερώτηση. Οπότε θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο βοήθεια στι τοπικέ αρχέ, γιατί τελικά αυτέ οι αρχέ επιζητούν το να υπάρχει μια ανθεκτική βιώσιμη λύση για τους πρόσφυγες. Έχω τώρα δύο ερωτηματάκια. Τελευταία. Το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή όσον αφορά τα θεσμικά όργανα ως προς τις ΜΚΟ, επιδεινώνεται. Έχουμε ένα σωρό δηλώσεις των πολιτικών φορέων, ακόμα και υπουργών κάποιων χώρων και από τη δική μου χώρα. Και με αυτές τις δηλώσεις θέτουν ένα αμφιβόλο τον ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα να αμφιβάλλω τις αληθείς προθέσεις, την ουδετερότητά τους όσον αφορά την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Αυτό είναι θέμα που θα πρέπει να το δούμε. Να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να ανασχέσουμε αυτή την τάση. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε μια χώρα που σίγουρα δεν είναι από τις πιο πλούσιες στην Ευρώπη και επιπλέον βρισκόταν ε, σε μια ε, κρίση, η οικονομική κρίση απασχόλησης, οπότε όπως γνωρίζετε οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ίδια κυβέρνηση ανέκαθεν αναγνώρισε ότι χωρίς την ευρωπαϊκή βοήθεια δεν θα μπορούσαν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Πάντως ο ρόλος των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά την ε, άμεση απόκριση σε αυτήν την κατάσταση ανάγκης ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Άρα δεν θα πρέπει να χάσουμε τη συμβολή αυτών των ΜΚΟ. Οπότε τα προβλήματα με τις ΜΚΟ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όλοι ξέρουμε ότι αν υπάρξει ένα εθνικό πρόγραμμα Τη ελληνική κυβέρνηση που θα εγκριθεί οι ΜΚΟ που θα κάνουν ό,τι τους έρχεται. Θα πρέπει να οργανώσουν ε, τη δραστηριότητά τους στα πλαίσια αυτού του εθνικού προγράμματο, βέβαια. Και όλοι γνωρίζουμε ότι γενικώ υπάρχουν προβλήματα αλλά θα πρέπει το μήνυμά μας να είναι διτό ότι είναι αναγκαίο οι ΜΚΟ να αναγνωριστούν όσον αφορά το έργο που έχουν επιτελέσει για αυτή την κατάσταση ανάγκες και αυτό το συμβούλιο που οργανώνεται να συνεργαστεί με την εθνική κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση ούτω ώστε να ξεκινήσει όταν εγκριθεί αυτό το εθνικό πρόγραμμα. Μίλτος Κύρκος, ευχαριστούμε Ενρικέ Μίλτο. Πες μας δύο λόγια για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ευχαριστούμε και την ΑΕΡΣΥ και η Λίντα και εγώ. Ήταν πολύ σημαντική η αποστολή που κάναμε. Being part of Greece, you are grateful for the Commission, for the mobilization. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ελλάδα είναι ευγνώμων ε, και για την αναγνώριση του προβλήματος ε, και για ε, τη συμφωνία με την Τουρκία που σταμάτησε τις ροές. Από την αρχή, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ο Κλόντ ήταν επικεφαλής της προσπάθειας αυτής, συζητούσαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν αμφισβητούμε τη θέληση της κυβέρνησης, ιδίως μετά την άφηξη του κ. Μουζάλα. Αλλά η διοικητική ικανότητα είναι αμφισβητήσιμη, γιατί η Επιτροπή απαιτεί να γίνουν τα κονδύλια αποδεκτά και να απορροφηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Αβραμόπουλος μας είπε την Άνοιξη ότι λιγότερο από 10% των κονδυλίων απορροφήθηκαν, άρα πρόβλημα υπάρχει. Και όσον αφορά την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των κονδυλίων, Όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει εικόνες ε, ανθρώπων που πεθαίνουν κατά από το που δεν είναι καθόλου η καλύτερη δυνατή εικόνα. Αλλά αυτά μπορούμε να τα αφήσουμε στο παρελθόν. Τα προβλήματα στην υπηρετική χώρα έχουν επιληθεί, βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες και μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να δουλεύουμε για την ένταξη των ε, ατόμων αυτών όταν θα αρχίσει να γίνεται η διαχείριση από το κράτος και όχι από την υπατιαρμοσία και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, θα πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση και αυτό είναι και το σωστό που πρέπει να γίνει, να αναλάβει τις ευθύνες το κράτος. Όμως, ε, ε, στη Μόρια, στη Λέσβο, μέχρι τα τέλη Μαΐου, οι γιατροί του κόσμου υποστηρίζαν τους γιατρούς. 10 γιατροί, 8, 11 νοσοκόμες, 8 ψυχολόγοι κλπ. Και τηλεφώνησα στο Υπουργείο και του είπα ότι μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι είναι οι γιατροί του κόσμου και το Υπουργείο μου είπε ότι ε, όντως αλλά η διαδικασία θα είναι 15 Αύγουστο και τίποτα δεν είναι στην Ελλάδα το 15 Αύγουστο, αλλά θα πάει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και ε, μας είπαν ότι είναι εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, άρα ο Ερυθρός Σταυρός ε, εξασφαλίζει καλές συνθήκες. Κάναμε όμως έρευνα και είδαμε ότι αντί των αριθμών που μας είχαν αναφέρει, ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρει δύο γιατρούς, ε, δύο νοσοκόμες και ένα ψυχολόγο. Και αντί 24 ώρες υποστήριξης, ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρει 8 ώρες την ημέρα υποστήριξη. Φοβόμαστε λοιπόν πάρα πολύ ότι η αλλαγή από το προηγούμενο καθεστώς στις υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος θα είναι καταστροφική. Και περιμένουμε κάποια απάντηση από την Επιτροπή. Γιατί σας ήταν τόσο δύσκολο να δημιουργήσετε ένα εθνικό σχέδιο ανταπόκρισης της ανάγκες που θα ήταν κοινό αποδεκτό. Να κάτσετε δηλαδή στο τραπέζι και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με το Μουζάλα και με τις, τους νέους φορείς που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εξασφάλιση των υπηρεσιών, γιατί αυτά τα τηλεφωνήματα που έκανα εγώ για να κάνω αυτή τη διερεύνηση θα πρέπει να έχουν γίνει οργανωμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρηματοδοτεί όλη αυτή την προσπάθεια, ούτω ώστε να μην, να μην υπάρχει κανένα κενό, γιατί ξέρετε ότι η κατάσταση στα νησιά είναι από, πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί συνεχίζει να υπάρχει κάποια ροή από την Τουρκία. Έχουμε γύρω στα 64 άτομα την ημέρα και συνεχίζουν έρχονται από την Τουρκία γιατί δεν λειτουργεί σωστά η συμφωνία με την Τουρκία 100% και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό και ξέρετε ότι προστίθενται άτομα στα στρατόπεδα. Χθε στη Μόρια κάηκαν πέντε ε, κοντέινερς και τρει μεγάλες σκηνέ. Πρέπει να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη του. Θέλω να ευχαριστήσω του Προέδρου και τη Επιτροπή ΝΤΕΒΕ και τη ΛΥΜΠΕ γιατί μα έδωσαν την ευκαιρία αυτή και ελπίζουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η ε, ελληνική πολιτική ηγεσία θα, θα μπορούσαν να ήταν σήμερα εδώ και ο κύριος Μουζάλης δυστυχώς είχαν ε, άλλες ε, υποχρεώσεις. Αλλά αυτά είναι προβλήματα που υπάρχουν από το 2015. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρέμβει ήδη από τον πρώτο χρόνο της κρίσης, το δεύτερο χρόνο της κρίσης, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους uh, τρεις θεσμούς και την ε, ΕΚΟ και ε, την τη HOME και την υπατιαρμοστία. Νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι εξαιρετική. Τώρα, πάρα πολλά χρήματα έχουν δοθεί, 400 εκατομμύρια. Ε, και άλλα 300, πολλά χρήματα. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σταθερότητα, χρειαζόμαστε βιωσιμότητα των δράσεών μας και πρέπει να δούμε ότι οι τομείς όπως η ένταξη, η προστασία των συνόδευτων ανηλίκων είναι προγράμματα που πρέπει να υλοποιηθούν. Και ε, δεν μπο... είναι απαράδεκτο να μιλάμε σήμερα για την κατάσταση στην Ελλάδα και να μην είναι εδώ αρμόδιος υπουργό και να μην είναι κανείς παρόν που θα εκπροσωπεί την Ελλάδα. Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το εθνικό πλάνο που υπάρχει, ποιο είναι το εθνικό σχέδιο. Πρέπει να το γνωρίζουμε και πρέπει και η Επιτροπή ε, να, ε, να το γνωρίζει. Επιτροπή ε, είναι πρόθυμη να επενδύει ε, σε αυτά τα προγράμματα βοήθειας, αλλά θα πρέπει και από ελληνική πλευρά να υπάρχει ανταπόκριση. Ακούσαμε ότι οι Δήμοι και οι κοινότητε φέρουν μεγάλο βάρος ε, και θα πρέπει και η Ελλάδα να είναι έτοιμη να απαντήσει στην Επιτροπή μας. Ποια είναι τα μέτρα για την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών, τι κάνουν με τους ασυνόδευτους ανηλίκους, πώς έρχονται από τα νησιά στην υπηρετική χώρα. Τι γίνεται με την ανακατανομή προσφύγων σε άλλες χώρες μέλη. Πώς μπορούμε να δούμε διαφορετικά την κατάσταση ε, με την Τουρκία και το θέμα των επιστροφών. Μετά την αλλαγή της κατάσταση στο Χαλέπι, Έχουμε μεγάλο αριθμό επιστροφών. Ελπίζω να υπάρχει, να συνεχίσει να υπάρχει βούληση επιστροφής στην πατρίδα. Πάντως, παρακαλώ τις ελληνικές αρχές να παρουσιάσουν το εθνικό πρόγραμμα δράσης, να μας το υποβάλουν και εμείς ως επιτροπές και ΛΥΜΠΕ και ε, ΔΕΒΕ θα πρέπει να είμαστε σε κατάσταση να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία η ελληνική κυβέρνηση μας παρουσιάζει. Πρόεδρος Μωράες. Ε, ε, είναι ο κύριο Βούλιο εδώ, εκ μέρου τη ελληνική πλευρά. Δεν θέλω να τον βάλω σε δύσκολη θέση. Θα μπορούσε στο τέλο να ε, μιλήσει, αν το επιθυμεί. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι τις 12 ε, και 4 στην Έχετε κι άλλο ένα σημείο που πρέπει να συζητήσετε μετά το τωρινό σημείο, οπότε δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Ο κύριος Χρυσόγωνος, παρακαλώ. Αν μπορείτε να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να διευκρινίσω κάποια ζητήματα που υπάρχουν παρανοήσεις. Υπόθηκε ότι η Ελλάδα έχει λάβει 500 εκατομμύρια ευρώ. Όμως αυτό είναι το συνολικό ποσό που έχει δοθεί στην Ελλάδα για το 2017 και για τα επόμενα δύο χρόνια. Από αυτό το ποσό, μόνο το 92% έχει λάβει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση έχει ξοδέψει περισσότερα από λίγο παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Από το συνολικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδόν τα μισά Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δοθούν ή να είχαν δοθεί για προστασία των συνόρων, άρα αυτό σημαίνει ότι ο αληθινός προϋπολογισμός για πολιτικές που ε, σκοπεύουν να βοηθήσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι ουσιαστικά το ίμιση του συνολικού ποσού. Σε κάθε περίπτωση. Αυτή τη στιγμή στα νησιά όπου η χρηματοδότηση περνάει από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο ελληνικό κράτος. Έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες για να ελαφρύνει το βάρος που φέρουν οι πρόσφυγες και μετανάστες. Ωστόσο δεν είναι καθόλου εύκολο το εγχείρημα και πρέπει να γίνει σταδιακά. Και σε ό,τι αφορά την υποδοχή κονδυλίων κεφαλαίων που έχουν ε, κατανεμηθεί, η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο περίπου τον, στο μέσο όρο των λοιπόν κρατών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το πολύ σημαντικό, δεδομένων των διαφόρων προαπαιτουμένων που υπάρχουν για να μπορεί η χώρα πραγματικά να πάρει, να λάβει αυτά τα κονδύλια, αυτά τα κεφάλαια. 40 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για λόγους που δεν έχουν να κάνουν άμεσα με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτό είναι ένα παράπονο που κατατίθεται, αλλά έχουν δοθεί για την ελληνική ακτοφυλακή έτσι ώστε να περιπολεί ε, για να σώσει ζωές στο Αιγαίο. Νομίζουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ για το σωστό σκόπο. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Χρυσόγωνε και για την ακρίβεια και για τη συντομία σας. Η, κυρία Λόπεθ Αγγιλάρ, ο κύριος Κώστα και στη συνέχεια αν ε, δεν διαφωνείτε να έχουμε τον εκπρόσωπο της ΜΕΑ που θα πάρει το λόγο της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο. Λίντα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις να θέσω από δική μου πλευράς. Να πω καταρχάς ότι Συναντήθηκα με τον Υπουργό Μουζάλα και με την μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία όταν επισκεφθήκαμε τα ελληνικά νησιά. Ήταν εξαιρετικά βοηθητικοί όλοι τους. Έχουμε δει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες βελτιώσεις που έχουν επέλθει σε σύγκριση με το παρελθόν. Όλοι το έχουν δει αυτό. Ε, δύο πράγματα με ανησυχούν. Jean-Luc Brugger, θα πάτε την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Θα συναντηθείτε και με μη κυβερνητικέ οργανώσει. γιατί πολλέ από αυτέ έρχονται και μα λένε ναι, ακούμε ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδο. Αλλά θα συναντήσετε, γιατί μπορούν να σας παρουσιάσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το που υπάρχουν κενά. Π.χ. μου είπαν ότι άκουσα ότι ναι, παρόλο που έχουν δημοσιευθεί π.χ. διαγωνισμοί, Υπάρχει κενό με το ποιος θα ε, είναι ο, ο, που θα έχει την εποπτεία, τη μέρημνα, την κηδαιμονία όταν θα αποσυρθεί η ΕΚΟ. Ίσως ε, πρέπει και οι δύο Γενικέ Διευθύνσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συναντηθούν και με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει να ακούσουν την πλευρά του. Και τι θα γίνει και τον ε, Αύγουστο, γιατί το είπε και ο Ενρίκε Γκερέρο, ότι κανεί δεν ξέρει ε, πότε θα και αν θα αποσυρθεί η Τουρκία από αυτή τη συμφωνία. Τα νέα δεν είναι καλά από την τουρκική πλευρά. Και όταν μιλούμε για την εκπαίδευση και την ε, ένταξη των παιδιών, προσφύγων παιδιών, των ανηλίκων, και την ενσωμάτωση, όπως είπε και το UNHCR. Τα παιδιά που είναι στους καταβλισμούς προσφύγων πηγαίνουν στο σχολείο το απόγευμα, μετά που έχουν τελειώσει τα ελληνόπουλα το σχολείο τους. Αναρωτιέμαι, η προσοχή δίδεται στην εκπαίδευση των παιδιών, στην σχολική φίτησή τους, γιατί οι οικογένειες με τις οποίες μελήσαμε στην Αθήνα που μένουν στους καταβλισμούς μας έλεγαν ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν και πολλά στα σχολεία. Είναι πολύ δύσκολο, άλλωστε ορισμένες και οικογένειες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα και αυτό πλέκει τα πράγματα. Τα παιδιά όμως πρέπει να πάνε στα mainstream σχολεία, τα κανονικά σχολεία και θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Ευχαριστούμε. Λίντα. Φερνάντο Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές και θλιβερό συνάμα το ότι έχουμε πάρα πολλούς και καλούς λόγους να συναντιόμαστε ξανά και ξανά για την ελληνική και ιταλική κατάσταση, για την ανθρωπιστική κρίση που σχετίζεται με την αποκαλούμενη προσφυγική κρίση. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι ο υπουργό κ. Μουζάλλας δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και θα ήθελα να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά, διότι είχα την πρόθεση να του απευθύνω διάφορες ερωτήσεις, διότι δεν υπάρχει μία, ένα λεπτομερές δημόσιο δημόσιο σχέδιο ανταπόκρισης και διαχείρισης της μεταβατικής της μεταβατικής ε, περίοδου ε, σε διαβούλευση με την ε, κοινωνία των πολιτών και λοιπούς φορείς. Θα ήθελα να είχα μπορέσει να θέσω ερωτήματα στον κύριο Μουζάλα για την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων στα σχέδια για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, γιατί αυτή είναι η πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Όμως, αφού είναι παρόντες εκπρόσωποι από τη Γενική Διεύθυνση Home και τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, θέλω να, τους, να στραφώ προς τα αυτούς, προς εκείνους και να τους ζητήσω να υπάρξουν τα συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστημάτα με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και τους εκπροσώπους των αρμοδίων αρχών και φορέων που θα αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα. Δεν υπάρχει δημόσιο σχέδιο αντιμετώπισης όλων αυτών διαθέσιμο. Είναι κρίσιμο αυτό το ζήτημα ότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχει σχέδιο συγκεκριμένο δημοσιευμένο για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση και μιλήσαμε για την απουσία, έχει γίνει λόγος για την απουσία πολιτικής βούλησης για τις δύο χώρες. Θα πρέπει να επιδειχθεί αλληλεγγύη. Άκουσα επανειλημμένος και θέλω να το θεωρήσω αξιοσημείωτο ότι για παράδειγμα η Ισπανία Πολλοί από εμά παραπονιόμαστε για την ε, συμπεριφορά τη ισπανική κυβέρνηση και για την έλλειψη επίδειξης αλληλεγγύης από πλευρά τη ισπανική κυβέρνηση, και αυτό πρέπει να το πούμε. Και ε, υπάρχουν κατηγορίε και ανάθεμα τα οποία πέφτουν πάνω στι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οποίε καλύπτουν το κενό που έχουν δημιουργήσει τα κράτη-μέλη που δεν έχουν πολιτική βούληση και ε, διαφάνεια και σαφήνεια. Ευχαριστώ. Ο κ. Κέστερ, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Υπάρχει και το θέμα της επανένωσης των οικογενειών ε, και ήθελα να θέσω αυτό το θέμα ε, για την επανένωση οικογενειών μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών μελών. Εκατοντάδες τον άσυλο ε, έχουν οικογένειες που βρίσκονται ήδη στη Γερμανία από ό,τι έχω πληροφορηθεί και σύμφωνα με τον κανονισμό του Βλήνο 3 υπάρχει δικαίωμα ε, επανένωση των οικογενειών. Σύμφωνα με τον κανονισμό, έχουν το δικαίωμα οι οικογένειες ε, στη διαδικασία αίτησης ασύλου ε, να κάνουν αίτηση στην ίδια, στο ίδιο κράτος μέλος όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Παρά αυτή τη νομικής απέτησης, αυτή η επανένωση των οικογενειών μέσω τη ε, αίτηση ασύλου στο ίδιο κράτος μέλος είναι περιορισμένη. Αυτό έχει αποφασιστεί από το Γερμανικό Υπουργείο. Και μόνο 70 άτομα το μήνα μπορούν να ε, έρθουν στην Γερμανία για τη διαδικασία της ασύλου. Δεν είναι αυτή μια διαδικασία αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και κατά πόσο αυτό αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υπάρχουν και αριθμητικά στοιχεία από το fact της Επιτροπής για τη διαχείριση των προσφύγων. Ένα ποσό 500 ευρώ που αναφέρεται Δεν ξέρω αν μπορούν οι εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων να μας πούν και εκπρόσωποι από την ΥΠΑΤΗ ε, αν μπορούν να μας πούν ε, τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε στους συναδέλφους. Ο κύριος ε, Βουλγαρίς νομίζω, αν μπορείτε να λάβετε το λόγο, δεν σας ζητώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά αν μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια από τα βασικά σημεία. Και βέβαια θα θέλαμε να μεταβιβάσετε κάποια από τα βασικά σημεία που αναφέρθηκαν σήμερα εδώ στον Υπουργό. Αν θέλετε, έχετε το λόγο για να αναφερθείτε σε κάποια από τα ερωτήματα που ετέθησαν σήμερα το πρωί. Έχετε δύο-τρία λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ και που μου δίνετε το λόγο. Συγγνώμη ειλικρινά που άργησα να έρθω, δεν ήμουν ε, ε, εδώ την αρχή της συζήτηση. Ο Υπουργός Μουζαλής βρίσκεται στην Ρώμη για διαβουλεύσεις με την Ιταλική κυβέρνηση, γιατί υπάρχει μια εξελισσόμενη κρίση στην Κεντρική Μεσογείο. Όλοι γνωρίζετε ότι τα πράγματα εκεί είναι πάρα πολύ κρίσιμα και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά. Γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τις ελληνικές αρχές, και από τον κύριο Μουζάλα και από όλους, για να αντιμετωπίσουμε ε, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό από το 2015 και μετά. Είχε την ευκαιρία ο κ. Μουζάλας και ευχαριστεί που μπόρεσε να συζητήσει με σας και επανειλημμένα. Ελπίζει θα μπορέσει να τα ξαναπείτε και πάλι με μεγάλη του χαρά για όλα αυτά. Επίσης ευχαριστούμε για όλη την βοήθεια που έχουμε δεχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα κράτη-μέλη και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πάντοτε συνεργαζόμαστε στενά και η πρόθεσή μας είναι να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Έλαβα υπόψη όλες τις παρατηρήσεις, όλες τις ανησυχίες, θα τις διαβιβάσω σε ελληνικές αρχές και θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Δύο μόνο την έχω να σας πω σαν ασυνόδευτος ανηλίκους. Ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Εμείς όλα ένα και περισσότερο. Βρίσκουμε κι άλλες, κι ε, λύσεις για να τους στεγάσουμε. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω της οικονομικής δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας για να καλύψουμε την παιδεία για όλα αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να πάνε στα σχολεία, με ειδικά προγράμματα. Προσπαθούμε επίσης να τα εμβολιάσουμε. Όλα αυτά είναι δύσκολα γιατί μιλούμε για μεγάλους αριθμούς. Πρόκειται επίσης για μεγάλους αριθμούς που πρόκειται να φιλοξενηθούν και στα άλλα κράτη-μέλη. Θα κάνει ό,τι μπορεί ο κύριος Μουζάλα, θα συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό το θέλουμε και προς χάρη των μεταναστών. Σας ευχαριστούμε, λέει κύριος Μωράς. Λίντα, δεν ξέρω, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έχουμε τρία λεπτά, δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω μήπως εσύ θέλεις για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Πρέπει να δώσουμε τον λόγο στην Επιτροπή, στον Σάιμον Μόργι, προσπαθήσω να σας καλύψω κάποια από αυτά τα οποία ελέγξαν πρώτα το γιατί τις ΜΚΟ που τα είπε ο κύριος ε, Γκερέρο Σαλόμ. Ναι, εκτιμούμε την προσπάθεια, το έχει το έργο τους. Είναι βασικό κομμάτι των προσπαθειών που κάναμε για τα προβλήματα της Ελλάδος και επαναλαμβάνω, δεν σταματάει η χρηματοδότηση προς τη ΜΚΟ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 100% εκτιμούν το ρόλο τους. Απλώς είπαμε ότι τώρα η οικονομική υποστήριξη θα έχει διάβλο το εθνικό πρόγραμμα. Το είπαμε αυτό στον ε, κύριο Μουζέλα. Εάν θεωρηθεί ότι χρειάζονται και άλλοι πόροι για την κρίση, πρόκειται να συμπληρώσουμε την οικονομική αυτή αρρωγή, ούτω ώστε να υπάρχει αυτή η ανταπόκριση ο πλευράς Ελλάδος για την κρίση. Στις 30 Ιουνίου είχαμε μια προσφορά για διαγωνισμό όσον αφορά στέγαση για τους ε, ε, ασύνοπτους ανηλίκους. Είχαμε πολλές προτάσεις από τις ΜΚΟ και τώρα αξιολογούνται αυτές. Ε, και ελπίζω τελικά να μπορούν κάποιες συμβάσεις μέχρι πρώτης ογδόου από πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Είπες για συνέχιση της προστασίας Λίντα όσον αφορά τους ανηλίκους και ακριβώς ο πλευράς Ελλάδος καταβάλλουν τώρα προσπάθειες όσον αφορά την μέρημνα και επιμέλεια αυτών. και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση οπότε και εμείς συνεχίζουμε με ευελιξία να καλύπτουμε τα κενά προσπαθούμε να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους ε, χρηματοδότηση ήδη για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση για τους ανηλίκους. Τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος ε, Κύρκος, είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ε, αρχές και, και όλη, όλη η υπηρεσία, η υπηρεσία του Ζουν Λουί, όλοι προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια ολική κάλυψη των οικονομικών αναγκών. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, ας δημοσιοποιήσει ό,τι θέλει η ελληνική πλευρά για αυτά Θέλουμε για το 2018 να αρχίσει τώρα η προσπάθεια προγραμματισμού για να μην έχουμε κανένα κενό. Να γίνουν όλα έφτακτα όπως προεπιτρώσουν όσον τους καταβλισμούς όπως σας έχει πει και ο κύριος Αβραμόπουλος. Φεβρουάριο του 2017 ήταν ε, η τελευταία επαφή μας και είπαμε ότι 1,8 εκατομμύρια έχουν ε, δοθεί για το άνευ και 4,2 ε, από το ISF. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, θα συνεχίζουμε να έρουμε όλα τα κενά, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει η περισσότερη Ελλάδα πέραν των όσων είπαμε ότι πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία της δήλωσης με την συνεχίζουμε και έχουμε αφήξεις 10.000 10.000 ε, κάθε βράδυ έρχονται και χάνονται πολλές ζωές και από τότε που ε, είχαμε τη συμφωνία με την Τουρκία, οι 10.000 γίναν 60. Παρ' όλα αυτά περισσότεροι φτάνουν ε, κάθε μέρα στην ε, Ελλάδα από όσους γυρίζουν στην Τουρκία. Και αυτό γιατί συνεχίζει να υπάρχει εμπλοκή όσον αφορά τη δεύτερη φάση των αιτήσεων ασυλουπία στη Μοριά πρόσφατα και είπα στον επικεφαλής του καπιταλισμού ήταν Χριστούγεννα, θέλετε να κάνετε μια ευχή. Τι θα ε, ε, είχατε ευχηθεί. Θα θέλαμε, είπε, επιτάχυνση της διαδικασίας. Ο κόσμος περιμένει πάρα πολύ χρόνο. Να, αυτό εξηγεί γιατί είχαμε αυτά τα προβλήματα στη Μόρια χθε. Άρα θα πρέπει επιγόντως να επιταχύνουμε τη δεύτερη φάση της διαδικασίας αίτησης ασύλου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας για να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές. Να υπάρχει ομαλή μετάβαση από τη διαχείριση της κρίσης σε κάποιο είδους βιώσιμη διαχείριση. Πολύ σύντομα θα είμαι. Όντω, ο ρόλο των τοπικών αρχών είναι κέριο και θα πρέπει να βελτιωθεί ο διάλογο μεταξύ κρατικών και περιφερειακών αρχών. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι παραμένει κάποιος φόβος από πλευρά ελληνικών αρχών όσον αφορά το τι θα γίνει με την ε, Συμφωνία ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκίας. Είχαμε μιλήσει με τον κύριο Μουζάλα και είχε συζητηθεί γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τα στρατόπεδα. Και ο λόγος ήταν ότι θέλουν να κρατήσουν ένα μαξιλάρι σε περίπτωση ε, που υπάρξει μια επιδείνωση της κατάστασης μεταξύ Ελλάδας ε, και Τουρκίας όπως περιέγραψε και ο Σάιμον πριν από λίγο. Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Έχουμε στην Ελλάδα 15 ε, εταίρους, οι 12 είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις και συμφωνώ ότι είναι σημαντικός ο ρόλος τους και Αναμπέλ στην ε, παρέμβασή της ε, το τόνισε. Ε, χρειάστηκε να δημιουργηθεί το πλαίσιο διαλόγου μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που είναι επαγγελματίες στην ανθρωπιστική βοήθεια αλλά δεν ήταν εξοικειωμένες με τον τρόπο λειτουργίας μιας κυβέρνησης Επομένω, έπρεπε να βρεθεί ο τρόπο συνεργασία και έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθώ και με μη κυβερνητικέ οργανώσει και θέλω να τονίσω ότι έχουμε συνεχή διάλογο. Ε, κάθε 15 μέρε έχουμε βίντεο ε, συναντήσει ε, με μη κυβερνητικέ οργανώσει και παρακολουθούμε πολύ στενά το τι γίνεται μέσω των υπηρεσιών μας επιτόπου και στα νησιά έχουμε τέσσερις ε, οργανώσεις εταίρους, είμαστε σε επαφή μαζί τους και είμαστε σε θέση να κάνουμε επακριβή αξιολόγηση για τα πιθανά κενά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ίσως να διαβάσατε ότι υπήρξε κάποιο περιστατικό στην είσοδο ε, ενό στρατοπέδου στην υπηρετική Ελλάδα ε, χθε και έγινε κάποια διαδήλωση στο στρατόπεδο. Μέσα σε λίγες ώρες βρήκαμε τι το προκάλεσε και τι έπρεπε να κάνουμε για να ανταποκριθούμε σε αυτή την κρίση, διότι υπάρχουν οι μα μας επιτόπου, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν άμεσα να συνομιλήσουν με τις ελληνικές αρχές και να βρεθεί κάποια λύση. Σα το ανέφερα σαν μεμονωμένο περιστατικό για να σα δείξω ότι υπάρχει λεπτομερέστατη παρακολούθηση από δική μα πλευρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα γίνει μια πολύ ομαλή μετάβαση και ο Αύγουστος θα είναι ένας ομαλός μήνας και θα δίδεται σε όλους ε, αυτό το οποίο πραγματικά τους αξίζει. Και όπως είπε και ο Σάιμον, έχουμε συνεχή διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ομιλητές. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Λίμπε, Ευχαριστώ τον Κλόντ και την Υποτιερμοσία. Και θα τα ξαναπούμε μετά το καλοκαι... τις καλοκαιρινές διακοπές θα συνεχίσουμε και κλεισμένων των θυρών για το επόμενο σημείο. Παρακαλώ λοιπόν να παραμείνουν μόνο ε, όσοι ασχολούνται με το θέμα αυτό για την Ερυθέα. Και παρακαλώ όσοι αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.